Καλημέρα σας, καλημέρα Επίτροπε, καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. Πρώτο θέμα είναι η έκθεση του κυρίου Βό, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Πριν δώσω ευθύς αμέσως τον λόγο στον εισηγητή, γνωρίζω ότι η εν λόγω συζήτηση, βέβαια όπως όλες, ε, είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση. Γι' αυτό θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να τηρήσουν το χρόνο αγόρευσης ε, για να μπορέσουμε στη διαδικασία προσέλκυσης προσοχής του Προέδρου Κατστιάη να δώσουμε το λόγο και σε όσους συναδέλφους έχουν εγγραφεί. Καταρχάς θα δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Φως για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Εκτός μικροφώνου, έχουμε να συστήσουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα πώς ε, στον ψηφιακό κόσμο μπορούμε να προστατεύσουμε τα πνευματικά δικαιώματα, πώς θέλουμε ε, να προσαρμόσουμε την κατάσταση, θέλουμε την πνευματική ιδιοκτησία να την προστατεύσουμε όσο μπορούμε και τα πνευματικά δικαιώματα μας ανήκουν, σε ποιον ανήκουν τέλος πάντων. Θέλουμε ένα νομικό πλαίσιο για το ίντερνετ ώστε ε, να μην υπάρχει κλοπή των έργων των δημιουργών. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που μας απασχολεί σήμερα και σε ποιο βαθμό θα πρέπει αυτά όλα να τα σταθμίσουμε και με τα θέματα που άπτονται της ελευθερίας, της έκφρασης και της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας. Περί αυτού πρόκειται. Στο ίντερνετ τελικά θέλουμε να τα αφήσουμε όλα ελεύθερα, να τα επιτρέπουμε όλα ή θέλουμε να υπάρχει προστασία και να ισχύουν κάποιες αρχές. Επίσης, πολλή συζήτηση γίνεται για το άρθρο 13 Πάρα πολλοί κόσμος εκεί εστιάζει. Θα ήθελα όμως ε, να ε, δώσω προσοχή και στο υπόλοιπο περιεχόμενο της οδηγίας. Ε, δηλαδή, ο στόχος μας είναι να έχουμε ένα σύγχρονο, μια σύγχρονη εξόριξη δεδομένων και κειμένων. Αυτό θέλουμε να εφαρμόσουμε, ώστε να είναι μια προοδευτική τεχνολογία και να προσφέρει όλες τις δυνατότητες που μπορεί. Ό,τι αφορά επίσης το άρθρο 12, ε, δίνουμε τη δυνατότητα ε, να υπάρχει και εδώ η δυνατότητα τα κράτη τα οποία πλήττονται να μπορούν να βρουν ε, μία ισορροπία σε ό,τι αφορά τους δημιουργούς και τους εκδότες βιβλίων, τους συγγραφείς δηλαδή και τους εκδότες. Επίσης για μικρούς καλλιτέχνε για το δημιουργικό κλάδο δηλαδή, για τους ηθοποιού κτλ. Έχουμε το άρθρο 14, ώστε και από εκεί και πέρα, δηλαδή όλα τα άρθρα μετά το 14 δίνουν τη δυνατότητα στο να υπάρξει μια καλύτερη σχέση μεταξύ των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων, ε, εκδοτών κτλ. Ε, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει συνέχεια κάποιος στο δικαστήριο. Βελτίωση δηλαδή της κατάστασης και εδώ. Επίσης με το άρθρο 11 δίνουμε τη δυνατότητα ε, για τους εκδότες ε, τύπου να έχουν μια καλύτερη προστασία και ουσιαστικά τους δίνουμε αυτό το δικαίωμα. Αυτοί θα δουν πώς θα το ε, χειριστούν, πώς θα το εκμεταλλευτούν. Όμως θέλουμε να είναι στην ίδια κατάσταση, να είναι ισότιμοι ε, με τους υπόλοιπους εκδοτές, διότι στο ίντερνετ, ε, επειδή η υπερτερή έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο τι γίνεται στο ίντερνετ, σε ό,τι αφορά τη δωρεάν δυνατότητα εκμετάλλευσης κάποιων έργων. Και δεν πρέπει πρέπει να τους αφήσουμε εκτός τους εκδότες. Αν δει κανεί το άρθρο 13... Ε, εμείς ε, έχουμε βρει και έναν ορισμό όπου γίνεται λόγος μόνο για ε, τις πλατφόρμες ε, που ξέρουν ακριβώς ότι χρησιμοποιούν την πνευματική ιδιοκτησία άλλων και κερδίζουν πολλά χρήματα. Στοχεύουμε ακριβώς σε αυτές το θέμα είναι βέβαια πώς θα εφαρμοστεί τεχνικά το μέτρο αυτό που οι πλατφόρμες καλούν ε, τους χρήστες να αναφορτώσουν ό,τι επιθυμούν ακριβώς. Θα, υπάρχει, θα πρέπει όμως να υπάρχει ευθύνη για τις ε, πλατφόρμες. Θα πρέπει να υπάρχει ευθύνη σωστής ε, χρήσης των δικαιωμάτων μας ιδιοκτησίας άλλων ή της πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Νομίζω ότι με τη δουλειά που κάναμε έχουμε μια πολύ καλή βάση, βάση της οποία μπορούν πλέον να δώσουν ε, τι οδηγίε του στα κρατημέλη για το πώ θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η οδηγία σε κάθε κράτο. Αυτό νομίζω ότι ήταν ο σωστό δρόμο, είναι ο σωστό δρόμο για να προχωρήσουμε προ τα επόμενα και να βρούμε την ισορροπία μεταξύ ελευθερία από ψηφιακού κόσμου και πνευματική ιδιοκτησία. Σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά, τον κύριο Ντάντι. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Οπωσδήποτε χρειάζεται αναθεώρηση του κοινοτικού πλαισίου για τα πνευματικά δικαιώματα. Η οδηγία καταδεικνύει ότι το Κοινοβούλιο πολλές φορές δέχτηκε αυτή την αρχή, ιδιαίτερα ως προς την εξισορρόπηση των πλατφορμών. Ο βομβαρδισμός ε, στην ψηφιακή αγορά δείχνει ότι προσπαθεί κανείς ε, να ξεφύγει από το πραγματικό περιεχόμενο. Δεν είμαστε υπέρ της λογοκρισίας. Θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει διάδοση πληροφοριών σε σχέση με κερδοσκοπικούς σκοπούς. Ως προς τις ψευδείς ειδήσει υπάρχουν αυτοί που θα ήθελαν το δίκτυο να είναι μια άγρια δύση των μεγάλων πλατφορμών. Όμως θέλουμε να ανταμείψουμε του, τα πνευματικά δικαιώματα και τους δημιουργούς που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος Γκάμπρι. Η Επίτροπος Γκάμπριελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητή, αγαπητέ εισηγητά, σκιώδης. Θα ήθελα τώρα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε τα τελευταία δυόμιση χρόνια η οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ψηφιακής αγοράς, της ενιαίας μας αγοράς αναγνωρίζουμε ότι μία προσωρινή πολιτική συμφωνία εξευρέθη για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Αγαπητά μέλη, πρόκειται για ένα ε, σημείο ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή πνευματική κληρονομιά και τις ευρωπαϊκές αξίες. Η νέα οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα μας επιτρέπει να φτάσουμε στους κοινού στόχους σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα του 21ου αιώνα η οδηγία τάσεται υπέρ εκείνων που προασπίζονται, που προασπίζουν τα πνευματικά δικαιώματα. Πρόκειται για τους εκδότες, παραγωγούς έργων, τις ψηφιακές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, συγγραφείς και ούτω καθεξής. Υπερασπίζεται τη δημιουργία και την τεχνητή ευφυΐα έτσι ώστε η πνευματική μας κληρονομιά να είναι πιο εύκολα προσβάσιμη στους πολίτες. Για πρώτη φορά στην ομοθέσια μας οι μεμονωμένοι πνευματικοί δημιουργοί θα ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους θέση και θα μπορούν να έχουν μία σωστή ανταμοιβή. Αγαπητά μέλη, όλοι αυτοί οι δημιουργοί αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει η πολιτιστική μας ε, κληρονομιά και η δημοκρατία μας. Αυτό ζητούν οι δημιουργοί. Θεωρούμε ότι το πλαίσιο αυτό είναι εξισορροπημένο αλλά και φιλόδοξο, έτσι ώστε οι δημιουργοί και όσοι κατέχουν πνευματικά δικαιώματα να μπορέσουν να ανταμείβονται σωστά. Οι πάροχοι υπηρεσιών επίσης θα ανταμείβονται όπως πρέπει καθώς και οι δημιουργοί γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε μία ανακοίνωση για την ε, ε, κατάσταση σε σχέση με την ε, μετάδοση αθλητικών γεγονότων και το κείμενο προσαρτάται στο, στην οδηγία νομοθετικού περιεχομένου, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αναμένω τις δικές σας, τη δική σας γνώμη και πιστεύω ότι με την υποστήριξη της οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα θα αποστείλουμε ένα στεναρό μήνυμα υπέρ των δημιουργών μας και των εν γέννη αξιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Για ένα λεπτό, ο κ. Κρασμετόρσκι από την Επιτροπή Ιτρέμ. κύριε Πρόεδρε. Η οδηγία είναι απαραίτητη. Το γνωρίζουμε όλοι. Όταν οι οδηγίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκαν πριν από καιρό, νομίζαμε ότι θα ήσχαν για πολύ καιρό. Και όμως ε, ήδη είναι πεπαλαιωμένε. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις διαβρώνουν, διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισμό Νομίζουμε ότι τα είχαμε κάνει όλα και όμως όχι. Το αντίθετο μάλιστα θα έλεγα, το διαδίκτυο είναι πεδίο μάχης για τους κολοσσούς της πληροφορίας με αποτέλεσμα να πιέζονται, να στριμώχονται στη γωνία δημιουργοί και ερμηνευτέ. οι οποίοι εν τέλει δεν αμείβονται για το έργο τους για να μην πω ότι είναι θύματα εκβιασμού. Επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι μουσείων, δημιουργοί, περιμένουν λύση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει ό,τι μπορεί, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναβάλουμε την απόφαση για την επόμενη ολομέλεια. Δεν είμαστε ακόμη όριμοι να πάρουμε απόφαση από την πολιτική Ζουλό. Κυρία Πρόεδρε, τα πλεονεκτήματα τα ανέφεραν άλλοι. Δεν θα τα επαναλάβω. Το ερώτημα είναι ένα. Τι σημαίνει αυτή η ψηφοφορία για την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει τη χαρά να είναι μπροστά στην ψηφιακή ρύθμιση και να αποτελεί υπόδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Θέλουμε πλειοψηφία είτε για να συνεχίσουμε να είμαστε στο προσκήνιο πρωτοπόροι, είτε για το αντίθετο. Η ψηφορία αφορά δυστυχώ το όλα ή τίποτα. Το θέμα είναι εάν ε, θα υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των μεν ή των δε. Εμείς θέλουμε να ωφελήσουμε τους πολίτες, τους δημιουργούς, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κόσμος θέλει ένα δίκαιο διαδίκτυο με ανοιχτέ πλατφόρμες όπου αμείβονται οι δημιουργοί και οι ερμηνευτέ, όπου προστατεύονται τα δικαιώματα. Αυτό ακριβώς λέει το κείμενο το οποίο ψηφίζουμε και η ψηφοφορία μας αφορά ένα θέμα. Οι πλατφόρμες έχουν ή όχι ευθύνη έναντι της κοινωνίας μας. Αυτό είναι το μόνο ερώτημα στο οποίο καλούμεθα να απαντήσουμε. Και νομίζω ότι όλη η Ευρώπη είναι υπέρ ολη η ευρωπη ειναι υπερ ενό ναι το Μπονί, από Το άρθρο 13 σε διάφορες αμφιβολίες από την αρχή, γι' αυτό χρειαζόμαστε και και χρειαζόμαστε μια συμβαστική λύση. Το διαδίκτυο δεν είναι απλώς η πρόσβαση σε διάσημους δημοσιογράφους. Είναι χώρος δημιουργίας, ψηφιακή δημιουργία μάλιστα και το χρησιμοποιούμε όλοι. Δεν μπορούμε να λέμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης. Πρέπει να ελέγχουμε και να ελέγχουμε και τα δικαιώματα. Εάν εσείς προωθείτε το προϊόν σας, το παστή ενδεχομένω, γιατί όχι. Και αυτό το αναγνωρίζει η μηχανή, το φίλτρο, οι πλατφόρμες. Και εκεί οι πλατφόρμες θα είναι προσεκτικές. Και ως προς το περιεχόμενο, ούτως ή άλλως, αποφασίζετε εσείς. Στο παρελθόν, υπήρχε η γνωστή σε όλους μας λογοκρισία. Σήμερα όμως αυτό είναι λάθος. Είμαι υπέρ της διαγραφής του 13 και τότε και μόνο τότε θα υπερψηφίσω μια κατά τα άλλα πολύ καλή οδηγία. Και συγχαρητήρια στον Άξελ με την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Συναδελφοί, ε, Σα άφησα λίγο περισσότερο χρόνο για τους εκπροσώπους των επιτροπών. Θα είμαι πιο αυστηρή από εδώ και πέρα. Σφόποντα. ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεταρρύθμιση του τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων για τους χρήστες, τον, για τις πλατφόρμες, για τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Και χαίρομαι που η πρόταση αυτή, η οδηγία αυτή, προστατεύει τα δικαιώματα των δημιουργών και την πολιτιστική κληρονομιά. Χαίρομαι που προστατεύονται έτσι τα δικαιώματα όσων δημοσιεύουν και κάνουμε και κάτι για τις πλατφόρμες που παρανόμως διαδίδουν περιεχόμενο. Δεν πρόκειται προφανώς για λογοκρισία. Η λογοκρισία στο διαδίκτυο θα ήταν κάτι διαφορετικό. Θα θα είχαμε λογοκρισία αν αποτρέπαμε δημιουργούς, δημιουργικούς ανθρώπους να κερδίσουν αξιοποιώντας το ταλέντο τους στο διαδίκτυο. Δεν θέλουμε να τους στείλουμε στην παρανομία ή σε μερική επασχόληση αφού πέρασουν μια μέρα οδηγώντας ταξί. Λοιπόν, χαίρομαι για το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου. Ήταν καλύτερο από ό,τι ανέμενα. Η κυρία Γκέριγκερ Έντενμπεργκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία δύο χρόνια συζητήσαμε διάφορες εκδόσεις του άρθρου 13 και τώρα καθίσταται σαφές ότι αυτό το κείμενο θα αλλάξει το διαδίκτυο όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα και θα υπάρχουν πολύ αρνητικοί αντίκτυποι στον ε, επιμερισμό της γνώσης. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους δημιουργούς, αλλά στο τέλος τέλος ε, δεν φτάνουμε σε μια σωστή εξισορρόπηση. Είναι μεγάλο σφάλμα. Άρα η μόνη μας επιλογή είναι να διαγράψουμε το άρθρο 13. Αυτός είναι απαράβατος όρος έτσι ώστε οι ψηφιακές επιχειρήσεις να μπορέσουν να δράσουν γιατί ήδη έχουν αντιδράσει σε αυτό το κείμενο. Η εντολή που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να υπερασπιστούμε τις ΜΜΕ από το άρθρο 13 Δυστυχώς όμως θα είναι αναγκασμένες να αγοράσουν ε, ακριβή τεχνολογία φιλτραρίσματος που διαθέτουν μόνο οι Αμερικανοί γίγαντες. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουν προσπάθειες για, οποιαδήποτε, ε, για οποιοδήποτε πλαίσιο αδειοδότησης. Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Υπάρχει μία μπλε κάρτα από τον κύριο Ρόντε. Κύριε Ρόντε, ίσως μπορείτε να ασχοληθείτε με το θέμα κατά το χρόνο μιλία σας. Ο κύριος Καρίμ για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ τον Άξελ για αυτή την εξαιρετική εργασία. Συνάδελφοι, η δική μου προτεραιότητα είναι να καταστήσω σαφές ότι οι δημιουργοί θα μπορούν να ζήσουν στα πλαίσια της άσκησης των δικαιωμάτων τους, ε, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας με το κοινό. Αυτό είναι αναγκαίο με βάση τα νέα μοντέλα και πλατφόρμες που υπάρχουν. Δεν ήταν εύκολη η διαπραγμάτευση, αλλά είμαι ικανοποιημένος γιατί φτάσαμε στους στόχους και υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Γι' αυτό θα υποστηρίξω την έκθεση κατά την ψηφοφορία γιατί έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις. Η εξόριξη δεδομένων θα είναι δυνατή για εμπορικούς σκοπούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά. Το άρθρο 11 βελτιώθηκε έτσι ώστε η βιομηχανία δημοσιεύσεων να είναι ασφαλής. Θα μιλάμε μόνο για μικρές εξορίξεις οι οποίες εξαιρούνται επιγραμμικά. Επίσης, ε, ε, δεν θα υπάρχει δυνατότητα εμπόρευσης των δεδομένων μέσα στα πλαίσια της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Και συνεχίζεται ο κατάλογος. Υπάρχει ευελιξία για τα κράτη-μέλη και δεν θα υπάρξει εποπτεία των χρηστών. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες πλατφόρμες πλατφόρμες προσπαθούν να πείσουν διαφορετικά το κοινό, στην ουσία το κοινοβούλιο ε, δεν θα δεχτεί αυτή τη ροπή πραγμάτων που προωθούν ορισμένες πλατφόρμες. Κύριε Ρόντε, διαδικαστικό. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Είναι παράλογο ότι αποτρέπεται τη δεξαγωγή συζήτηση. Μας βλέπει σήμερα όλο ο κόσμο και έρχονται όλοι εδώ στην Ολομέλεια για να διαβάσουν τον λόγο που φτιάξαν στο σπίτι τους, αλλά συζήτηση δεν έχουμε. Αλλά το θέμα παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εσείς αποτρέπετε αυτή τη συζήτηση. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι σόφρον, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι δίκαιο. Συγγνώμη, Πρόεδρος. Συμφωνώ. Θα ήθελα να δώσω σε όλους χρόνο αγόρευσης. Δυστυχώ όμω υπάρχουν κάποιοι που θέλουν το λόγο και δεν είναι στον κατάλογο. Εσείς είστε στον κατάλογο και εγώ θα πρέπει να ιεραρχήσω ε, και θα δώσω το λόγο και στου συναδέλφου στη διάρκεια τη ε, διαδικασία Catch the Eye. Δεν μπορώ όμω να δημιουργήσω πρόβλημα με τις υπηρεσίε. Ε, δεν μπορώ να δώσω σε όλους το λόγο. Ελπίζω όταν σα δώσω το λόγο να μπορέσετε να πείτε αυτά που θέλετε. Σημειώνω όμω την παρατηρήσή σα. Ο κύριο Καβαντά για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί για πρώτη φορά σε μια Ήπειρο μια κοινοβουλευτική συνέλευση προσπαθεί να επανεξισορροπήσει τις σχέσεις μεταξύ γκάφα, αυτών των μεγάλων ομίλων και αυτών που τις τροφοδοτούν, δηλαδή δημιουργούσε και τύπο η δημιουργική κλάδη 130 δις ε, το χρόνο και 1.700.000 εργαζόμενοι στην Ευρώπη απειλείται από τις άδικους συσχετισμούς, τους οικονομικούς. Κάτι όμως ακόμα πιο επικίνδυνο, όσο όχι τόσο άμεσα, είναι ότι καταραίει ο τύπος, ε, η σχετική βιομηχανία και κανένας δεν προσπάθησε να το σταματήσει αυτό. Ο τύπος, κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είναι η βάση της δημοκρατίας. Όταν δεν θα έχουμε πλέον ελεύθερο τύπο, όταν δεν θα υπάρχει στο Google κανένας δημοσιογράφος, ούτε στο YouTube, ούτε στη Wikipedia, ούτε πουθενά άλλου, δεν θα έχουμε πλέον ενημέρωση, απλά μόνο φήμες σαν αυτές που ακούμε και κυκλοφορούν εδώ και ορισμένους μήνες. Αυτό το κείμενο είναι η μόνη ευκαιρία για τους δημιουργούς και για τις επιχειρήσεις του τύπου και τους Ευρωπαίους δημοσιογράφους να πάνε να εξισορροπήσουν προς όφελός τους και θα έλεγα να προστατεύσουν το μέλλον τους εξού και πρέπει να ψηφίσουμε το κείμενο και να το ψηφίσουμε συνολικά αρνούμενοι να δεχτούμε οποιαδήποτε τροπολογία. Το κείμενο αυτό πρέπει να το δούμε ως ένα πρόβλημα πρώτο βήμα, γιατί για να υπάρχει εξισορρόπηση στην όλη κατάσταση χρειάζονται και άλλα βήματα. Γίνεται λόγο για λογοκρισία, για φιλτράρισμα, ε, για τη Wikipedia μα μιλάνε, η οποία προστατεύεται στο κείμενο. Δεν υπάρχει λογοκρισία. Δεν υπάρχει φιλτράρισμα. Γιατί όμως φτάσαν μέχρι εδώ στην Ολομέλεια αυτές οι ιδέες, γιατί για πρώτη φορά μέσα σε 15 χρόνια που είμαι ευρωβουλευτής μας βομβάρδισαν σαν να είμαστε πολιτικοί κρατούμενοι, διανοούμενοι ε, τα ιερά τέρατα ε, της οικονομίας που θέλουν τις δραστηριότητες μας να τις φετεριστούν. Πρέπει να το ψηφίσουμε όλο αυτό το κείμενο συνολικά, γιατί αλλιώς ε, θα, αυτό θα έχει πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις διακόπτη το μιλητής.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 έχω ήδη στον κατάλογο και για το κατσέ και αυξάνει το αριθμό αυτό. Κύριε Ρέντε, τρεπτά κυρίε και κύριοι, τρία πράγματα σε αυτή τη συζήτηση που άπτεται των πνευματικών διωμάτων είναι πρωτοφανή. Πρώτα απ' όλα, 200.000 άνθρωποι αυτό το Σαββατοκύριακο διαδήλωσαν κατά τη μεταρρύθμιση αυτή. 5 εκατομμύρια έχουν υπογράψει ένα petition κατά του upload filter, του φίλτρου αναφόρτωση όμως ε, ε, δεν το έχει λάβει κανεί υπόψη, ότι ε, πρώτη φορά γίνεται τέτοια αναστάτωση κατά μιας οδηγίας της Ένωσης και αγνοείται εντελώς αυτή η διαμαρτυρία. Αντί όμως να υπάρχει κάποια κριτική, προσβάλλονται όσοι προσπαθούν να υψώσουν τη φωνή τους και έχουμε Όπω ίσως και ο κύριος Καβαντά πιστεύει, πολλού να θεωρούν ότι τα email δεν τα στέλνουν οι εκλογείς στους βουλευτέ, αλλά bots. Και η Κομισιόν λέει ότι είναι μία μάζα οι, ε, αυτοί που ασκούν κριτική. Και του Τσέντε, ο υπεύθυνο θεωρεί ότι πληρώνονται αυτοί που ε, διαμαρτύρονται. Ε, όλα αυτά είναι δυσφήμιση που πολύ εύκολα μπορεί κανείς να την αντικρούσει και θεωρούν κάποιοι ε, ότι ε, τέλος πάντων αυτά τα έχουν ξεκινήσει κάποιες ομάδες λόμπι και τα παρουσιάζουν ε, οι επιφυλίδες κάποιων εφημερίδων. Ε, θεωρούν ότι όλα αυτά κάποιοι προέρχονται από την Αμερική και έτσι δεν σκέφτονται επί της ουσίας ε, τι γίνεται. Δεν τους νοιάζει ε, που υπάρχουν προειδοποίησεις και από τον ίδιο τον Ομοσπονδιακό Υπεύθυνο για την Προστασία Δεδομένων σε ό,τι αφορά το upload filter και ο εκπρόσωπος για τα ελευθερία του ισαγνώμισε και πολύ σημαντικά ερευνητικά κέντρα για άλλα όματα. Κανένας δεν θεωρεί ότι είναι σημαντική αυτή η μεταρρύθμιση τσέντε ούτε τεσπεντέ ούτε και αντιπολίτευση ε, και κανείς δεν θέλει να πάρει την πολιτική ευθύνη για το upload filter του άρθρου 13 όπου το θεωρούν όλοι κάτι ανόητο μέχρι και η κυρία Μέλκε παρακαλώ λοιπόν να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας παρακαλώ διακόπτω γιατί θέλω να ερεμήσουν κάποιοι συνάδελφοι που φωνασκούν Κύριε Μπροκ, Παρακαλώ. Έχει το λόγο η κυρία Ρέντα αυτή τη στιγμή. Να σεβόμαστε παρακαλώ τον ομιλητή που είναι στο μικρόφωνο. Κυρία Ρέντα, συνεχίστε. Κανείς δεν θέλει να πάρει την ευθύνη ε, στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση ε, για το upload filter παρόλα αυτά ε, ψηφίζουν ε, στην ε, κυβέρνηση υπέρ και μάλιστα η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung έχει ανακαλύψει το ότι υπήρξε ένα παζάρ μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας δέχτηκαν οι Γάλλοι το upload filter για να ψηφίσει το Nord Stream η Γαλλία. Το πιο τραγικό, συγγνώμη λέει η πρόεδρος, Χαίρομαι που έχετε ξυπνήσει όλοι έτσι πολύ καλά σήμερα το πρωί. Παρακαλώ μην ακούτε από δεξιά από αριστερά φωνές. Το τραγικότερο είναι ότι η νέα γενιά που για πρώτη φορά θα ψηφίσει φέτος στις ευρωεκλογέ ήδη μαθαίνει το μάθημά της. Δηλαδή τους λέμε δεν αξίζει τίποτα η διαμαρτυρία σας, οι πολιτικοί θα συνεχίσουν να ψεύδονται και δεν θα επηρεαστούν καθόλου ούτε από τα πραγματικά στοιχεία και τα επιχειρήματα αν ε, αυτά δεν προωθούν τα γεωπολιτικά του συμφέροντα. Αυτό, η αίσθηση αυτή της αδυναμίας θα τους στιγματίσει τους νέους μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να προχωράμε γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την ελευθερία του διαδικτύου αλλά και μια ολόκληρη γενιά θα τους ε, ε, κλέψουμε αν θέλετε την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική και δεν είναι αυτό. Διακόπτεται η πρόεδρος. Πρέπει να καταψηφίσουμε το 13 λέει η κυρία. Ρέντα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κασπάρη έχει μια ερώτηση. Το δέχεστε? Το ερώτημα, ναι, το δέχομαι. Αξιότιμη συνάδελφε Ρέντα, ουσιαστικά ε, εμένα είπατε ότι είπα πως ε, είναι πληρωμένοι αυτοί που διαδηλώνουν. Να σας επαναλάβω ότι είπα ξεκάθαρα και σας παρακαλώ να ε, λαμβάνετε υπόψη αυτά που λέω εγώ και όχι αυτά τα οποία επίτηδε παρερμηνεύετε εσύ και η ΟΜΗ. Είπα εγώ ότι γίνεται δημοσία προσπάθεια ακόμη και με πληρωμένου διαλωτέ ε, να ε, μην προωθηθεί αυτή η οδηγία για την προστασία των Εγώ δεν μίλησα για του νέου για τι δισεκατομμύρια νέου και νέε οι οποίοι κατεβαίνουν. Διακόπτεται. Zeitung in einem Artikel mit der Über Κύριε Κασπάρη, 30 δευτερόλεπτα είχατε για να κάνετε μία ερώτηση. Αυτό που θέλετε να πείτε το είπατε. 30 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι ο κανόνα. Και έτσι λειτουργούμε, με κανόνε εδώ. Κυρία Ρέντα θα απαντήσει τώρα. Κυρία Κασπάρη, μόνο σας ε, το είπατε ότι κάποιοι διαδελτέ ήταν πληρωμένοι και μιλήσατε για 450 ευρώ. Σας ακούσαμε, σας ακούσαμε όλοι, είπατε για 450 ευρώ και ε, το για τα, ε, δικαιο, οργανισμός για τα δικαιώματα έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται εδώ ε, για να ε, έχουν επαφές άσκησης πίεσης. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όμως που πληρώνουν εδώ μόνοι τους τα τα οδηπορικά του. Θέλατε για διαδικαστικό κάποιο το λόγο. Λοιπόν, ένα λεπτό ε, έχετε χρόνο αγόρευση στη συνέχεια. Θέλετε τώρα μήπω να το χρησιμοποιήσετε το λεπτό σα. Εκτό μικροφώνου κάποιο φωνασκεί. Okay. Λοιπόν, παρακαλώ. Δεν με αφήνετε, φωνάζει κάποιο, να υποβάλω ερώτηση. Ψεύδεται η συνάδελφο, ψεύδεται ενώπιον τη ολομελία. Πρόεδρο, σα ακούω, αλλά δεν σα ακούν οι άλλοι, γιατί το μικρόφωνο σα δεν λειτουργεί. Κύριε Ρέντε, παρακαλώ, καθίστε. Εγώ ω πρόεδρο, θα φροντίσω όσοι προσήλθαν να έχουν χρόνο στο ΚΑΤΣΤΙΑΗ Αλλά δεν μπορείτε να διακόπτετε την συνεδρίαση. Κύριε Ρέντα, θα δεχτείτε μία σύντομη ερώτηση του κύριο Ρέντε. Ωραία, 30 δευτερόλεπτα κύριε, 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Σα ερωτώ λοιπόν, πού είναι το περίφημο φίλτρο αναφόρτωση. Πού είναι κυρία Ρέντα αυτό το upload filter συγκεκριμένα στο κείμενο. Πείτε μας πού είναι, πού το λέει. Έχετε 30 δευτερόλεπτα. με ρόντε, λέει ότι οι πλατφόρμες ε, θα πρέπει να ε, μην επιτρέπουν ε, την αναφόρτωση κατοχυρωμένων πραγματικά δικαιώματα και δεν χρειάζεται να έχουν κάποια άδεια. Και λέει εκεί ότι μπορούν να έχουν αυτό το upload filter, αυτό το φίλτρο, να γίνεται αυτό το φιλτράρισμα αναφόρτωσης. Please, Παρακαλώ, συνάδελφοι. Κύριε Μαστάλκα, 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή συνεδρίαση μοιάζει μάλλον με τελικό παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου. Δεν μοιάζει με κοινοβουλευτική συνεδρίαση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μιλώ εξ όλων αν ε, έλεγα ότι θα είμαστε όλοι ανακουφισμένοι όταν υπερψηφιστεί το κείμενο. Αλλά και αν δεν ψηφιστεί, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Έχουμε τα άρθρα 11 και 13, τα πιο επίμαχα, τα πιο αμφιλεγόμενα. Κοιτάξτε, μετά από ένα μισό χρόνο δεν είμαι ευχαριστημένο με το αποτέλεσμα. Εγώ θα είμαι κατά τη πρόταση. Πάντω, σπαταλήσαμε μια εξαιρετική ευκαιρία να εξυγχρονίσουμε τον χώρο τη πνευματική ιδιοκτησία και να υποστηρίξουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ανταυτού, έχουμε μια πρόταση η οποία εξαπαρά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εισάγει λογοκρισία, ευνοεί τα chat και εν τέλει ευνοεί τα μέσα κοινωνική δικτύωσης. Θα είναι το τέλος του διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε. Μπορώ να αναφέρω πολλά παραδείγματα, αλλά δυστυχώ δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Επιπλέον πιστεύω ότι εάν υπερψηφίσουμε τη σημερινή έκθεση, αυτό θα είναι χαστούκι στο πρόσωπο εκατομμυρίων ανθρώπων που μας στέλνουν ε, email ε, και διαμαρτύρονται στους δρόμους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, πρέπει να κάνει κάτι για να μην χάσει την αξιοπιστία του. Τέλος πια στην υπεροψία. Να έρθουμε πιο κοντά στους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά, Μας πιέζουν και δύο πλευρές. Από τη μια πλευρά ακούμε για χιλιάδες ανθρώπων που ανησυχούν για το μέλλον του ίντερνετ και από την άλλη έχουμε ακριβέ δεξιώσει ε, υπέρ του κειμένου. Μην νομίζετε πάντως ότι οι δημιουργοί στηρίζουν την πρόταση. Οι μεγάλοι παίκτε την υποστηρίζουν. Εμένα όμως με ενδιαφέρουν οι ψηφοφόροι μου, οι απλοί άνθρωποι, οι καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την πολυτέλεια να χρησιμοποιούν λόμπιστ. Ε, Τι χρειαζόμαστε, μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δημιουργών και από την άλλη μεριά ε, της προστασίας των καθημερινών απλών ανθρώπων. Η προτινόμενη νομοθεσία, ειδικά με τα άρθρα 11 και 13, δεν πετυχαίνει αυτήν την ισορροπία. Πρόκειται για ανελεύθερο μέτρο, διότι στην πράξη οι μεγάλες εταιρείε θα χρησιμοποιούν τους πολίτες ως ε, αυτομάτως ενόχους. Θα σταματήσει το περιεχόμενο να αφαιρείται αυτομάτως. Έτσι, ισοπεδώνοντας τα πάντα, γνωρούμε τους εθνικούς κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δυστυχώς δεν υπάρχει μία λύση για όλα. Πρόκειται για ναρκοπαίδιο. Εν τέλει, το νόμιμο περιεχόμενο θα αντιμετωπίζεται ως παράνομο. Τι βλέπω λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον, η γνώμη των Βρετανών που θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αλλάξει. Και όσο και το αντίθετο. Πού πηγαίνουμε. Φοβούμαι ότι κάποιοι που ήταν υπέρ της παραμονής τώρα θα ψηφίσουν Brexit λόγω αυτής της νομοθεσίας. Λοιπόν, με την πρόταση αυτή απομακρύνουμε τους νέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κακή νομοθεσία. Είναι δυστυχώς νομοθεσία της τελευταίας στιγμής. μετά από τρει μισή εβδομάδε εμεί θα έχουμε κλείσει την ε, θητεία μα. Λοιπόν, α μην βιαστούμε για άλλη μια φορά. Δυστυχώ δεν λάβαμε υπόψη μα αυτά που έπρεπε να λάβουμε υπόψη μα. Ακούστε, αφουγκραστείτε του ψηφοφόρου σα. Α έρθουμε πιο κοντά στον Βρετανικό λαό, στο λαό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μπλε κάρτα. Το κύριο Στρογεύσκη, την δέχεστε. 30 δευτερόλεπτα. Είμαι ένας από τους τελευταίους ε, που συντάσσονται με τα λόμπι, όμως θα ήθελα να ξεχωρίσουμε τα διαφορετικά λόμπι. Κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αγώνα για το δικαίωμά τους στην αμοιβή. Η ερώτησή μου προς σας, κυρία, είναι δεν βλέπετε ότι υπάρχουν τα μεγάλα εμπορικά λόμπι οι γίγαντες της αγοράς και οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι απλώς διεκδικούν την αμοιβή τους. Ευχαριστώ. Καμία αντίρρηση. Να αμείβονται αυτοί που πρέπει να αμείβονται. Και καλώς υπεραμείνονται του δικαιώματός τους. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, επαναλαμβάνω. Καμία αντίρρηση. Όμως, ξανά και ξανά τη βλέπουμε τα μεγάλα συμφέροντα, αυτά που μας πιέζουν, παρά οι δημιουργοί. Οι δημιουργοί στη δική μου εκλογική περιφέρεια λένε ότι δεν τους ακούμε. Αν και εν τέλει κανείς δεν θέλει αυτή την νομοθεσία. Οι απλοί πολίτες ανησυχούν με το άρθρο 11 και 13. Πρόεδρος, και από τον ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Σήμερα ε, ασχολούμαστε με την οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι μία ιστορική ημέρα ή μία μαύρη ημέρα αντίθετα. Είναι απότοκη ε, τριετούς εργασίας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση ίσα-ίσα ε, σφετερίστηκε το όλο ζήτημα η Silicon Valley. Δεν υπερασπιζόμαστε τους δημιουργούς και χρήστες. Οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιγραμμικές ε, πλατφόρμες που πολλές φορές αποσύρουν το περιεχόμενο. Οι δημιουργοί έχουν δικαίωμα ίσης και δίκαιης αμοιβή. Ο Μαλρό έλεγε ότι ότι ο πολιτισμός δεν κληρονομείται, κατακτάται. Ο Σκιώδης λοιπόν λέω ναι στον πολιτισμό, ναι στα δικαιώματα των δημιουργών, των εκδοτών και των καλλιτεχνών. Ο κύριος Φουντούλης για ένα λεπτό. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και ειδικά στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζουν λογοκρισία βασισμένη αποκλειστικά στις επιθυμίες και τα συμφέροντα των ιδιοκτητών τους. πώς άραγε νομιμοποιούνται οι ιδιωτικοί φορείς να περιορίζουν θεμελιώδεις ελευθερίες; οι σημάνσεις και η κατηγοριοποίηση του περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο στιγματισμού ή εξοβελισμού ανεπιθύμητων ή ανταγωνιστικών ιδεών και προσώπων. για παράδειγμα μόνο η απλή αναφορά του ονόματός μου ή κοινοποίηση ομιλία μου στην ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου σε συγκεκριμένο μέσο κοινωνική δικτύωση, αρκεί ώστε να τιμωρηθεί ο κάτοχο του λογαριασμού με ποινή αποκλεισμού για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα ή να του κλείσουν το προφίλ. εάν λοιπόν σε αυτό το ήδη ζωφερό για την ελευθερία του λόγου περιβάλλον προσθέσουμε και οργουελικής εμπνεύσεω λογισμικά που θα ανοιχνεύουν τι απαγορευμένε λέξει. καταλαβαίνουμε πω θέτουμε τι βάσει για μια καταπίεση των ελευθεριών βγαλμένη από τι πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας που αρμόζουν μόνο σε σοβιετικά καθεστώτα. σας ερωτώ λοιπόν αυτό είναι το μέλλον που επιθυμείτε για την ένωση; εμείς σίγουρα όχι και γι' αυτό θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη έκθεση και κυρίως τη συγκεκριμένη διάταξη. ευχαριστώ. Η κυρία Φερχάιν για 1,5 λεπτό. Αξιότιμοι συνάδελφοι, εδώ και πάνω από δυόμιση χρόνια στο Κοινοβούλιο τσακωνόμαστε με τα κράτη-μέλη για να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη συμβιβαστική πρόταση. Και έχουμε ένα κείμενο επιτέλου ε, που θα οδηγήσει σε περισσότερη δικαιοσύνη στο διαδίκτυο και θα αναλάβουν τι ευθύνε του και οι μεγάλοι όμιλοι. Σίγουρα είναι δικαίωμα βασικό η προστασία των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. Ε, θέλουμε λοιπόν ε, να προστατευτούν τα έργα των δημιουργών. Η κοινωνία μας ε, δεν έχει στόχο ε, να μην προστατεύουμε. Θέλουμε κατά ε, ελάχιστα εισοδήματα και άλλα βασικά δικαιώματα. Δεν μπορούμε να βάζουμε, να μην βάλουμε εμπόδια στους μεγάλους ομίλους για να ζητάνε αστρονομικά ποσά και να κερδοσκοπούν σε βάρος των δημιουργών. Έχουμε λοιπόν πιο απλές διαδικασίες αδειοδότησης στο 70, το 17, στο 7, στο 9 ε, θέλουμε την κατοχήρωση της ελευθερίας έκφρασης. Υπήρχαν κάποιες δυσανάλογες διατάξεις, ε, τις οποίες ε, τις έχουμε απαλείψει. Dropbox, eBay, ε, Wikipedia δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία και επίσης ρυθμίζουμε τα όσα ισχύουν για τους μικρούς εκδότες και για τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι αναλογικά λοιπόν τα μέτρα και θέλουμε δικαιοσύνη στο διαδίκτυο. Οι πλατφόρμες είναι αυτές οι οι οποίες ε, ε, έχουν το περισσότερο κέρδος. Εμείς θέλουμε δικαιοσύνη, δεν θέλουμε άναρχο καπιταλισμό όπως αυτός που βιώνουμε εδώ. Θέλουμε ένα τέλος σε αυτόν τον άναρχο καπιταλισμό. For one minute, Madam Η κυρία Ροζιέρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η οδηγία είναι απότοκη μιας εργασίας δυόμιση ετών. Δημιουργεί εκδότες, δημοσιογράφοι, ερευνητές ε, έχουν συμμετάσχει, αλλά και οι ίδιοι οι καταναλωτές είναι άμεσα εμπλεκόμενοι, οι ίδιοι οι χρήστες γιατί θα μας δώσει την ασφάλεια δικαίου που θέλουμε και δεν θα είναι αυθαίρετες πια οι πλατφόρμες. Έτσι η Ευρώπη ε, θα μπορέσει να είναι κυρίαρχη σε σχέση με τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις που λαιλατούν τα προσωπικά δεδομένα, την ιδιωτική μας ζωή και καταπατούν τα δικαιώματα των δημιουργών. Πώς ε, είναι δυνατόν να μην αμείβεται η εργασία γιατί είναι σε ψηφιακό πλαίσιο. Όλοι πρέπει να αμείβονται. Τα μεγάλα ε, λόμπι ψεύδονται. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τις παραβιάσεις διαφάνειας και πολλές φορές υπάρχει σκιώδης χρηματοδότηση πλατφόρμων. Ελπίζω λοιπόν να σταθούμε κατά του άκρα του νεοφιλελευθερισμού και υπέρ των Ευρωπαίων Χριστών. Ο κύριος Λοσλοτόφσκι για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, μερικά χρόνια πριν ε, έγινε ε, μία, υπήρξε μία διχογνωμία για το τι μας απασχολεί εδώ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της οδηγίας είναι το γεγονός ότι η ερμηνεία θα είναι πιο σοβαρό ζήτημα από το ίδιο το κείμενο. Ο κύριος Βός δεν μας έπεισε με την παρουσίασή του. Δυστυχώς οι ορισμοί δεν είναι συγκεκριμένοι ε, και γι' αυτό ακριβώς θα υπάρξουν πολλά κενά και στη δημόσια συζήτηση. Δυστυχώς οι κολοσσοί ορίζουν τη δημόσια συζήτηση και τη μονοπολούν. Και γι' αυτό θα ήθελα να καταψηφίσετε αυτή την οδηγία. Ρόντε για ένα λεπτό. Κύριε, κύριε Ρόντε. Πραγματικά είναι απίστευτο το ότι εδώ σήμερα ακούμε Ε, την αριστερά να λέει πράγματα που κανονικά δεν λέει ε, η αριστερά. Ε, δεν υπάρχει, για να καταρρέψω, καταρρύψω κάποιους μύθους, δεν υπάρχει αναφορά στο upload filter. Δεν υπάρχουν φίλτρα αναφόρτωσης, ούτε περιορίζονται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Αντιθέτως, ελέγχεται κάπως η κατάσταση με τις πλατφόρμες το facebook και άλλοι γιγαντές δεχόμαστε σήμερα πολύ ε, ελαφρά την καρδία ε, να επηρεάζουν το τι μπορεί και το τι δεν μπορεί ε, να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ενώ οι δημιουργοί δεν έχουν ούτε δικαιώματα ούτε ελέγχουν τα δικά τους ουσιαστικά δημιουργήματα. Και Πραγματικά αυτή η κολοσσοί της τεχνολογίας που δεν πληρώνουν μισθούς, που δεν πληρώνουν φόρους, είναι ανεξέλεγκτοι. Και έτσι φτωχαίνουμε και οικονομικά και πολιτισμικά. Ελπίζω να στηρίξετε σήμερα το... Κυρία Τρούπελ έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλουμε ελεύθερο αλλά και επιτέλους δίκαιο ίντερνετ. Δεν θέλουμε ανευθυνότητα. Δεν θέλουμε όμως ούτε και λογοκρισία. Ε, στην Κίνα υπάρξει, υπάρχει λοκρισία, δεν υπάρχει προστασία πνευματικής συντοξίας. Αυτό που θέλουμε είναι οι ενεργές ε, πλατφόρμες περιεχομένου να έχουν άδεια ε, και έτσι θα είναι όλοι κερδισμένοι. Αυτός που θα αναφορτώνει θα έχει κάποια δικαιώματα και οι πλατφόρμες θα παίρνουν την ευθύνη επιτέλους και θα υπάρχει και μια αναλογική αμοιβή για το δημιουργό. Αυτό θα φέρει δικαιοσύνη στο ελεύθερο διαδίκτυο, κάτι που όλοι επιθυμούμε. Χρειάζονται γενικοί κανόνε ε, για τον καπιταλισμό των πλατφορμών. Πρέπει να πληρώνουν φόρου και να αναλαμβάνουν ευθύνε ε, όταν κάνουν ε, εκστρατεία πληροφόρηση. Θέλουμε την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας ε, και δεν μιλάμε για υπερίθμιση εδώ, αλλά για δίκαιους κανόνες, γιατί ε, είναι οι ε, κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων η μειοψηφία στην κοινωνία μας και χρειάζονται την προστασία μας. Ψηφίστε παρακαλώ το κείμενο αυτό, γιατί θα φέρει μεγαλύτερη δικαιοσύνη στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, κυρία Μίχελς. Βλέπω να χαιρετίζεται ορισμένη την εναρμόνιση ε, στα πνευματικά δικαιώματα. Όμως αυτοί που είναι υπέρ αυτής της μεταρρύθμισης ε, ε, λένε ότι ενισχύεται ο δημιουργικός κλάδος 5 εκατομμύρια άνθρωποι όμως και σας παρακαλώ και αυτοί είναι δημιουργοί, έχουν υπογράψει αυτή την αναφορά. Δεν θα πρέπει να παίρνουν αποφάσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα οι μηχανές. Γι' αυτό υπάρχει το κράτος δικαίου και αυτό το ε, άρθρο 13 ή 17 ε, γίνεται λόγος για αυτό το upload filter. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει αυτή η διάταξη για τις αδειοδοτήσεις. Ε, η ρύθμιση των πλατφορμών πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Ψηφιακό φόρο, ηθική αλγόριθμη, έλεγχος των καρτέλ ε, και καταπολέμηση των μονοπωλίων. Ας βρούμε λοιπόν καλύτερες λύσεις γιατί ουσιαστικά θέλουμε να έχουμε ελεύθερη επικοινωνία τον 21ο αιώνα και όχι εκαθάριση στο διαδίκτυο ότι δεν μας αρέσει. Mr. Patton, one minute. Against fair copyright. Είμαστε υπέρ της προστασίας των δημιουργών. Η οδηγία δυστυχώς προάγει τα συμφέροντα των πολυεθνικών, αυξάνει τα κέρδη τους. Έχει σκοπό να καταπνίξει τον ελεύθερο λόγο τη διαφορετική άποψη. Αυτό θέλουν τα καθεστώτα. Οι διαφορετικές φωνές ήδη αποκλείονται από τις πλατφόρμες. Αυτό κάνουμε ακριβώς με την οδηγία. Θεσμοθετούμε την λογοκρισία. Επ' αυτού ψηφίζουμε. Οι βουλευτές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι έχουμε σύντομα εκλογές. Οι ψηφοφόροι να σημειώσουν ποιοι υπερψήφισαν και ποιοι καταψήφισαν αυτήν την οδηγία και να καταψηφίσουν αντιστοίχως τον Μάιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μαζί με τους μεγάλους παίκτες να καταπνίξουν τις ελεύθερες φωνές. Ε, αυτοί οι βουλευτές που θα υπερψηφίσουν αξίζει να χάσουν τη θέση τους στο Κοινοβούλιο. Σώσουνε ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, χάρη στη συνεισφορά όλων, το διαδίκτυο είναι μια μικρογραφία του κόσμου μας. Σας ενοχλεί. Δεν θέλουμε υπερβολική νομοθέτηση. Το διαδίκτυο είναι το τελευταίο προπύργιο ελευθερίας και γι' αυτό κάποιοι δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Αυτό δείχνει ότι οι κανόνες σας είναι βλαβεροί θα μας ήταν καλύτεροι χωρίς αυτούς τους κανόνες. Αυτό είναι το διαδίκτυο, ελευθερία. Χωρίς τους κανόνες αυτούς θα είχαμε μια καλύτερη ζωή. Αυτήν προσπαθείτε να καταστρέψετε. Όποτε και όπως μπορείτε. Λοιπόν, όχι, δεν θα σας αφήσουμε να θέσετε τροχοπέδι στη ζωή, την ελεύθερη ζωή των ανθρώπων. Δεν θέλουμε τις παγίδες που προσπαθείτε να δημιουργήσετε στο διαδίκτυο. Πέδρος. κράντες Πασκουάλ για ένα λεπτό. Το περίφημο άρθρο 13 προσπαθεί να δώσει απαντήσεις για το τι θα κάνουν οι πλατφόρμες τη στιγμή που δεν προασπίζονται τα δικαιώματα των ε, δημιουργών. Και αυτό αφορά και τον τελικό χρήστη. Δηλαδή, ε, το περιεχόμενο θα πρέπει να την χάνει προστασίες, γιατί την πνευματική ιδιοκτησία την κατέχουν οι δημιουργοί, είτε είναι υλικό είτε άϊλο. Θα πρέπει λοιπόν να υπερασπιζόμαστε το περιεχόμενο των δημιουργών. Υπάρχει πνευματικό, πνευματική δημιουργία, γιατί η πλατφόρμα είναι αυτή που ευεργετείται από το περιεχόμενο μέσω διαφημίσεων. Η πλατφόρμα θα πρέπει να έχει την αδειοδότηση έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να καταλυστεύει το περιεχόμενο χωρίς ε, τη θετική γνώμη των δημιουργών. Αυτό ακριβώς είπαμε και στους τριμερείς ε, διαλόγους. Νομίζω ότι θα πρέπει να τύχει της υποστήριξής μας αυτή η προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέλκιν για ένα λεπτό. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Μόνο η Google είναι κατά τη μεταρρύθμισης, λένε αυτοί που είναι υπέρ τη οδηγία. Δεν ισχύει όμως αυτό. Ε, και ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μάλλον για τα προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και πολλοί άλλοι θεωρούν ότι τελικά ε, οι ε, φορείς διαχείρισης θα ισχυροποιηθούν. Όχι όμως οι δημιουργοί, γιατί τελικά πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από την πνευματική δοξία, αλλά με τη δημοκρατία μας έχει να κάνει. 5 εκατομμύρια υπογράφουν αυτή την petition και τους λένε ότι είναι ένα, μια μάζα ε, από την Κομισιόνα ε, και πολλοί ε, θεωρούν ότι αυτοί οι οποίοι είναι κατά δεν εκφράζουν τις γνώμες τους αλλά το έκαναν κάποια bot, κάποιες μηχανές το ε, διαδίκτυο ή ότι κάποιοι για να κατέβουν ε, στο δρόμο να διαδηλώσουν έχουν πάρει 450 ευρώ. Επομένως πλήττεται τη δημοκρατία μας. Πρέπει ιδίω τους νέους Ευρωπαίους να τους λάβουμε σοβαρά υπόψη οι οποίοι θέλουν ε, να παραμείνει το ίντερνετ όπως το θέλουν γιατί με το άρθρο το 13 και με το κείμενο αυτό καταστρέφεται το διαδίκτυο όπως το θέλουν. Πρέπει λοιπόν να διαγράψουμε το άρθρο 13. Ευχαριστώ. Κύριε Βέλκεν, έχετε από τον κύριο Ράτκε Μία μπλε κάρτα. Ναι, αγαπητέ ε, συνάδελφοι, ε, μα είπες ε, πώς οι άλλοι εκτός του Google είναι κατά η υπουργό δικαιοσύνη, η κυρία Μπάλα από το S5 δεν ήταν μεταξύ αυτών που αναφέρατε. Την ξεχάσατε. Ψήφισε στο Συμβούλιο υπέρα, αλλά τώρα λέει όχι πρέπει να ψηφίσουμε κατά. Άρα δεν τα έχουμε πολύ καταλάβει. Μήπω πρέπει να μα εξηγήσετε τι συμβαίνει. Αγαπητέ Ντένις, ε, τιμή μου να σε βοηθήσω να καταλάβεις. Ε, η ε, υπουργό δικαιοσύνη ε, ήταν κατά και ουσιαστικά έπρεπε να τηρήσει τη συμφωνία μεταξύ Μέρκελ και Γαλλίας που κατήγγειλε χθε η ΕΦΑΤΣΕΤ. Αυτό είναι ο λόγος λοιπόν. Ο κύριος Λούκε για ένα λεπτό έχει το λόγο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 Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πραγματικά ε, είναι απίστευτο αυτό το οποίο αποκάλυψε η ΦΑΤΣ, ε, η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Γίνονται παζαρέματα από τη μία το upload filter και από την άλλη ο Nord Stream. Ε, δεν είναι έτσι η πολιτική όμως. Κανονικά θέλουμε αντικειμενικότητα. Πρέπει να δούμε αν χρειάζεται τελικά αυτό το φιλτράρισμα για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής θυξίας. Κανείς δεν θέλει να στερήσει το εισόδημά τους από τους δημιουργούς. Τι κάνουμε όμως με αυτά τα φίλτρα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Και αν θεωρούμε ε, και λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχει αναφορά σε αυτά τα φίλτρα, σε αυτό το κείμενο, αυτό είναι αναλυθές. Πριν ε, δημοσιοποιήσουν το περιεχόμενο, οι πλατφόρμες πρέπει να έχουν ε, πρώτα επαληθεύσει κατά πόσο υπάρχει ε, ενδεχόμενο παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι φίλτερο. Είναι δηλαδή απλό filter μέσα στην ε, ε, οδηγία ε, και υπάρχουν κάποιοι μικροί ε, φορείς εδώ οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Το άρθρο 13 πρέπει να διαγραφεί από την οδηγία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ψηφίσουμε για την προστασία των δικαιωμάτων της Ευχαριστώ για να πει κυρία Τούμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συναδελφοί. Το ότι χρειάστηκαν μισή χρόνια για αυτήν την οδηγία δεν την κάνει δυστυχώ καλύτερη. Οι επιπτώσει στα δικαιώματα του ανθρώπου είναι πολύ σοβαρέ και το λένε πανεπιστημιακοί, ΜΚΟ, καθώ και ο ειδικό ε, για τα δικαιώματα του ανθρώπου από τον Ιωάννη Βασίλειο. Αν διαβάσουμε την ε, Οικουμενική Διακήρυξη, όλοι έχουν δικαίωμα στην πληροφορία μέσω οποιοδήποτε καναλιού, φορέα κλπ. Και αυτό ακριβώς καταργούν τα άρθρα 11 και 13. Δημιουργούν εμπόδια στην κυκλοφορία της πληροφορίας. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των δημιουργών. Ναι, όμως ε, εκεί έχουμε πολύ διαφορετικούς παίκτες. Δεν είναι ισόρροπη η πρόταση. Δυστυχώς εδώ βάζουμε μπροστά τα συμφέροντα των λίγων. Τον Σεπτέμβριο είχαμε πολλές εναλλακτικέ μπροστά μας στο τραπέζι και σήμερα όχι πια δυστυχώς. Οπότε θα καταργήσουμε τα 11 και 13 ή θα καταψηφίσουμε. Γιατί αλλιώ το πλήγμα κατά των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άντερσον, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δύο λόγια για την γελία θεωρία συνωμοσία του λόμπι του copyright. Εμείς θέλουμε ένα ελεύθερο διαδίκτυο Δεν θέλουμε να πέσουμε στην παγίδα του Google και του Facebook. Συγγνώμη, η θεωρία συνωμοσία είναι για τα σκουπίδια. Δίνουμε μάχη κατά αυτών των γιγάντων εδώ και χρόνια. Δίνουμε μάχη για την ιδιωτικότητα, δίνουμε μάχη κατά των μονοπωλίων. Εγώ θα ήθελα να χτυπήσουμε την Google και το Facebook εκεί που τους πονάει να, ψηφίσουν, να πληρώσουν φόρους Γι' αυτό να δώσουμε αγώνα. Να δώσουμε αγώνα για την ιδιωτικότητα, να δώσουμε μάχη για την ανάληψη ευθύνη. Όμω, εδώ πρόκειται για τη λάθο μάχη. Εγώ δεν εμπιστεύομαι το Google και το Facebook, αλλά εμπιστεύομαι του ειδικού που λένε ότι τα άρθρα 11 και 13 είναι κάκα για το διαδίκτυο και ότι δεν πρέπει να πέσουν θύματα αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Κύριο Κυρία Πρόεδρε, είναι καιρός να νομοθετήσουμε για να περιορίσουμε τους γίγαντες της Βορειοαμερικής, να βάλουμε ένα φρένο, να πληρώσουν αυτοί οι μεγάλοι τους δημιουργούς. Κατανοώ τις πιέσεις των γιγάντων του κλάδου, όπως το υπενθύμισε ο κύριος Καβαντά. Μιλάμε για 536 δισεκατομμύρια το χρόνο.